Good morning Καλημέρα σε όσους παρακολουθούν. Um, Θα σας δώσω το λόγο άμεσα στους ε, πράσινους, τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο, για να συζητήσουμε τα θέματα δημοσιονομικού ενδιαφέροντος. Για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, την κρίση και τις επιπτώσεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ε, είναι μέσα στην υποχρέωση, είναι μέσα στο ρόλο ενός Ευρωβουλευτή να δίνει το λόγο σε, στους πολίτες και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Ζούμε μια βαθιά κρίση στην Ελλάδα, είναι αλήθεια αυτό. Χρειάζονται αλλαγέ, αλλά αλλαγέ αυτέ πρέπει να είναι ισορροπημένε, δίκαιε και να είναι με τη συμμετοχή αυτών που θα υποστούν τι αλλαγέ. Αυτό σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε σίγουρα να είναι καλύτερο, Όλοι νομίζω θέλουμε ένα καλύτερο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από διάλογο, μέσα από τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών και όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, γιατί έτσι μπορούν να προκύψουν βιώσιμες και ουσιαστικές λύσεις. Ε, μάλλον δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν οριζόντια μέτρα, μέτρα τα οποία δεν είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει με ένα αρθρολογικό σχεδιασμό και αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε εδώ σήμερα με τη συμμετοχή ανθρώπων από τα πανεπιστήμια, των ε, ανθρώπων που ξέρουν ακριβώς τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, τι επιπτώσεις έχουν οι αλλαγές και στο χώρο του πανεπιστημίου, αλλά θα έλεγα και γενικότερα στην κοινωνία. Είναι μια εποχή που χρειάζεται να γίνουν βαθύτερες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία και αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν παρά και με τη συμμετοχή του πανεπιστημίου ως καταλήτη αυτών των αλλαγών αν χρειαζόμαστε κοινωνική καινοτομία, αν χρειαζόμαστε οικολογική καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία, αν χρειαζόμαστε νέες αξίες, νέες προτάσεις για την εξέλιξη κοινωνίας, αυτές δεν μπορούν να προέλθουν χωρίς τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη διέξοδο από αυτή την κρίση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εάν πλήτεται το Πανεπιστήμιο, σημαίνει ότι πλήτεται και ένας από τους θεσμούς ή ένα από, από τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να βγούμε από αυτή την κρίση πολύ περισσότερο όταν το Πανεπιστήμιο και η κοινωνία θα έπρεπε να προγραμματίζει για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ε, η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαδικασία, αλλά και πώς μπορεί να γίνει καλύτερη προετοιμασία προετοιμασία επομενης επόμενης προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Τόσο για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το ρόλο που θα παίξει το Πανεπιστήμιο για το Πανεπιστήμιο, αλλά και για το ρόλο που μπορεί να παίξει το Πανεπιστήμιο στο να εξελιχθούν η ε, οικονομική, να εξελιχθούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή, στην απασχόληση, στην προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμα και για τα προγράμματα όπως είναι τα ερευνητικά προγράμματα, το, το Horizon 2020, αλλά και πολλά άλλα, το Πανεπιστήμιο πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Και ακόμα περισσότερο όταν σήμερα συζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και στι διάφορε επιτροπέ και στην Ολομέλεια για την αναγνώριση των ισχυρών χαρακτηριστικών κάθε περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφώσει το δικό της μοντέλο ανάπτυξης, ο ρόλος του Πανεπιστήμιου σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντικός, ώστε να βοηθήσει και τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία των πολιτών, αλλά και τις περιφέρειες, στο να διαμορφώσουν μια νέα στρατηγική για την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία, και βέβαια στο να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν όλες αυτές τι κατευθύνσεις. Και δεν νομούμε μόνο μια εξεζητημένη έρευνα, αλλά και μια έρευνα που αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κοινωνικά, οικονομικά, παραγωγικά κάθε περιφέρειας. Αν λοιπόν την ίδια στιγμή πλήττεται το Πανεπιστήμιο και προσπαθεί να διασώσει τη λειτουργία του, τότε δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στους ανθρώπους από το Πανεπιστήμιο που ήρθαν ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσουν για το Πανεπιστήμιο, να ενημερώσουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη και τα πανεπιστήμια σε άλλες χώρες. Ήδη υπάρχουν ε, μηνύματα και από άλλους πανεπιστημιακούς και πανεπιστήμια θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο καταρχή στου πανεπιστημιακού. Σε λίγο θα είναι μαζί μα και η Ρεμπέκα Χάρμ, που είναι συμπρόεδρο τη ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα, έχει και, θα κάνει και αυτή μια σύντομη παρέμβαση. Στι 11 η ώρα θα υπάρχει μια ενημερωτική εκδήλωση ανοιχτή σε όποιον θέλει να την παρακολουθήσει. Θα είναι στην αίθουσα PHS 7C50 και σίγουρα θα έχουμε και άλλε παρεμβάσει Μου προσκληθεί και οι Έλληνε Ευρωβουλευτέ, αλλά και άλλοι φορεί. Ε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την ε, Βούλα Τσέτσι που είναι η Γενική Γραμματέας της Ομάδας των Πράσινων. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο. Σίγουρα ορισμένοι πανεπιστημιακοί είναι και ευρωβουλευτέ εδώ, αλλά νομίζω ότι δεν αφορά μόνο του πανεπιστημιακούς, δεν αφορά μόνο του ευρωβουλευτέ, είναι μια υπόθεση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, που είναι ο πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και είναι προεδρεύον τη Συνόδου των Πριτάνων. Και μετά θα, έχει, θα πάρει το λόγο ο κύριο Πάρη Τσάρτα, καθηγητή που είναι πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλο του Προεδρείου τη Συνόδου, καθώ και η καθηγήτρια η κυρία Ελένη Καραμολέγκου, που είναι πρόεδρο του Τμήματο Φιλολογία Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλο τη Πανεπιστημιακή Συγκλήτου. Ε, το λόγο στον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο Καλημέρα σας. Εκ μέρους της Συνόδου των Πριτάνεων θα ήθελα των ελληνικών πανεπιστημίων θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Ευρωβουλευτή, τον ε, Νίκο τον Χρυσόγελο για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας έδωσε να παρουσιάσουμε εδώ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο τα προβλήματα που ταλανίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και ιδίω το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό αυτό της διαθεσιμότητας ε, του διοικητικού προσωπικού οκτώ πανεπιστημίων. Ε, να ξεκινήσω από εκεί που άφησε τον ήμο ο κ. Χρυσόγελος. Πράγματι, η παιδεία είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, μοχλός ανάπτυξης, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή πλήττεται από την οικονομική κρίση. Η παραγωγή και η μετάδοση της επιστημονικής γνώσης αποτελούν σημαντικά συστατικά της οικονομικής ανάπτυξης και του δρόμου προς την κοινωνική ευημερία Επιπλέον, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα λειτουργήσε και ως ο σημαντικότερος μοχλός αναδιανομής, εισοδήματος και αναδιάταξης των κοινωνικών τάξεων, μια και ήταν αυτός ο θεσμός ο οποίος επέτρεψε παιδιά από αγροτικές ή φτωχές οικογένειες μέσω της πανεπιστημιακής τους μόρφωσης να γίνουν γιατροί, να γίνουν μηχανικοί, να γίνουν δικηγόροι, να γίνουν γεωπόνοι και έτσι να αλλάξει και η κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα αλλά και να ενισχυθεί ο δρόμος προς την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην παιδεία και στην ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο συγκεκριμένα, και ενώ θα περίμενε δηλαδή κανείς εν μέσω μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και ανάγκης αλλαγών στη χώρα μας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να αντιμετωπίσουμε την ύφεση και να ξαναμπούμε σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης, ενώ λοιπόν σε αυτό το σκηνικό θα περίμενε κανείς η παιδεία να αποτελεί τον βασικό μοχλό πάνω στον οποίο η πολιτεία θα έπρεπε να στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας, με λύπη του διαπιστώνει κανείς ότι η παιδεία είναι ένα ακόμη από τα θύματα της λιτότητας στον δρόμο της χώρας να αποκαταστήσει την, την οικονομική της κατάσταση. Ε, αντιμετωπίζεται δηλαδή η παιδεία σαν ένα τομέας ο οποίος μπορεί να συμβάλλει μέσω της λιτότητας, άρα μέσω της συρρήκνωσής του, ότι μπορεί να συμβάλλει στα δημοσιονομικά προβλήματα και στις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στους δανειστές της. Αυτό όπως αντιλαμβάνεται κανείς είναι μια πολιτική επιλογή. Θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι αυτό το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα εδώ, το θέμα της διαθεσιμότητας δηλαδή του διοικητικού προσωπικού στα πανεπιστήμια δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Τρόικα. Είναι πολιτική επιλογή της χειμερινή κυβέρνησης της Ελλάδας να πλήξει το διοικητικό προσωπικό των ελληνικών πανεπιστημίων. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει εάν πίστευε ότι τα πανεπιστήμια, η παιδεία είναι σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα στα, στην παιδεία στην Ελλάδα και ειδικά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εδώ και Τρία είναι ο τέταρτος χρόνος όπου τα πανεπιστήμια πληρώνουν το τίμημα της λιτότητας. Η πρώτη, το πρώτο, η πρώτη ένδειξη αυτής της κατάστασης ε, συνέβη με την δραστική μείωση των κρατικών προϋπολογισμών των ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι προϋπολογισμοί σήμερα βρίσκονται περίπου στο 40% αυτού που ήταν πρώτου 2010. Άρα υπήρξε μια μείωση στα τέσσερα αυτά χρόνια που μεσολάβησαν στους κρατικούς προϋπολογισμούς της τάξης του 60% και φέτος ανακοινώθηκε μια περαιτέρω μείωση της τάξης του 15% για τη νέα χρονιά, για το 2014. Δηλαδή Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μια τέτοια μείωση θα έπρεπε να έχει ακολουθηθεί και από μια μείωση του φυσικού αντικειμένου των πανεπιστημίων, εφόσον ο στόχος, όπως αποκαλύπτεται είναι η συρρήκνωση των πανεπιστημίων. Αυτό δεν έχει συμβεί. Κάθε χρόνο δια της μεθόδου της διολυστήσεως αυξάνουν οι φοιτητέ των πανεπιστημίων, αυξάνουν οι εισαγόμενοι στα ελληνικά πανεπιστήμια και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εξίσωση, η οποία μάλλον με ανίσωση μοιάζει παρά με εξίσωση, από τη μια μεριά αυξανόμενο φυσικό αντικείμενο για τα πανεπιστήμια, αυξανόμενο εκπαιδευτικό έργο, αυξανόμενο ερευνητικό έργο και από την άλλη μεριά δραστική συρρήκνωση των μέσων και των πόρων με τα οποία αυτό πρέπει να επιτελεστεί. Εάν ήταν μόνο το οικονομικό πρόβλημα, ε, θα σας έλεγα ότι αυτό έχουμε βρει τρόπους και το έχουμε αντιμετωπίσει. Έχουμε βρει τρόπους και έχουμε κάνει δραστική εξοικονόμηση των δαπανών των ελληνικών πανεπιστημίων. Έχουμε βρει τρόπους και έχουμε προσαρμόσει τις ανάγκες μας στα νέα οικονομικά δεδομένα. Και αυτό αν έχει συμβεί, έχει συμβεί σε αυτό που συχνά αποκαλούμε χάρη στον πατριωτισμό των ανθρώπων του Πανεπιστημίου, οι οποίοι με ελάχιστα μέσα οι ίδιοι προσωπικά λόγω της μείωσης και των δικών τους οικονομικών απολαβών, κυρίως όμως χωρίς μέσα που το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να τους διαθέτει, εφόσον ε, έχουν υποστεί δραματική μείωση οι, οι δημόσιοι προπολογισμοί των πανεπιστημίων. Εν εξακολουθούν και επιτελούν πάρα πολύ υψηλό έργο και όπως όλοι θα γνωρίζετε τα ελληνικά πανεπιστήμια σε όλες τις τελευταίες αξιολογήσεις παρά το γεγονός της μείωσης της δημόσιας χρηματοδότησης που ε, απολαμβάνουν εν βρίσκονται στα κορυφαία 1 με 2, 2,5%, 3% του συνόλου των πανεπιστημίων τα οποία αξιολογούνται. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι στο 0,98, είναι στο 1%. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι στο 1,2% ε, των πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο της, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο βρίσκεται στο 0, ε, είναι στο 1,96%. Όλα τα πανεπιστήμια τη χώρα είναι στο 1 με 2, 2,5% του συνόλου των πανεπιστημίων, σύμφωνα με τι πιο πρόσφατε αξιολογήσει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μάλλον καλά κάνουμε τη δουλειά μα, παρά το γεγονό των δραματικών περικοπών ε, στι δαπάνε μα. Δεν ήταν όμω μόνο οι οικονομικέ περικοπέ αυτέ οι οποίε χτύπησαν τα ελληνικά πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια. Από το 2010 και μετά, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό το οποίο για οποιοδήποτε λόγο έφευγε από το Πανεπιστήμιο, είτε λόγω συνταξιοδότηση κυρίω, είτε για άλλου λόγου, δεν αντικαθίσταται πλέον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για κάθε θέση η οποία εγκαταλείπεται και ενώνεται, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αντικατάσταση. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι υπήρξε μια δραστική μείωση και του προσωπικού τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπου ειδικά στο διδακτικό προσωπικό αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό, διότι όταν φεύγει ένας καθηγητής, σε ένα τμήμα, σε μια σχολή, αντιλαμβάνεστε ότι το γνωστικό του αντικείμενο δεν μπορεί να διδαχθεί από κάποιον άλλον. Υπάρχει λοιπόν και ένα πρόβλημα μείωση προσωπικού αυτή τη στιγμή στα ελληνικά πανεπιστήμια, το οποίο σε συνδυασμό με το οικονομικό ζήτημα ενισχύει τη δύσκολη κατάσταση. Όμω, εδώ, σε αυτό το σημείο, ενώ δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια κινούνται μεταξύ υποχρηματοδότηση και μείωση του προσωπικού, έρχεται η πολιτική τη διαθυσιμότητα από πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση η οποία επέλεξε να συμπεριλάβει στην διαθεσιμότητα και τα ελληνικά πανεπιστήμια, να δώσει το οριστικό χτύπημα, θα έλεγε κανείς, το τελειωτικό χτύπημα στα πανεπιστήμια. Με έναν τρόπο παντελώς αυθαίρετο, χωρίς καμία αξιολόγηση των διοικητικών δομών, μάλλον σε αντίθεση με την αξιολόγηση των διοικητικών δομών την οποία κάναν τα πανεπιστήμια και έβγαλαν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά στα οποία κατέληξε η κυβέρνηση, Καταφέρετο λοιπόν ατεκμηρίωτο και χωρίς αξιολόγηση τρόπο, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι στα οκτώ πανεπιστήμια της χώρας, τα οποία πλήττονται, υπάρχουν 1.349 διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι πλεονάζουν, οι οποίοι περισσεύουν. Εδώ θα πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Υπουργείου της Παιδείας μέσα στο καλοκαίρι, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να εφαρμόσουν μια ένα σχέδιο αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης των διοικητικών τους δομών. Πράγματι προχωρήσαμε σε αυτό το σχέδιο και αυτά τα σχέδια της αξιολόγησης των δομών μας, τα οποία στείλαμε στο Υπουργείο, απεδείκνυαν ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια χρειάζονται 2.500 ακόμα θέσεις διοικητικών υπαλλήλων προκειμένου να αποκαταστήσουν τα κενά τους και όχι 1.400 πλεονάζοντες όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση χωρί να δημοσιοποιήσει και χωρί να εξηγήσει, άρα έχουμε και ένα θέμα αδιαφάνεια εδώ, με ποιο τρόπο, με ποια μέθοδο, με ποια κριτήρια απέρριψε την αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστημίων, προχώρησε στην οριζόντια α, α, θέση σε διαθεσιμότητα 1.349 διοικητικών υπαλλήλων, χωρίς να εξηγήσει, χωρίς να δημοσιοποιήσει τη μέθοδο, τα κριτήρια της αξιολόγησης, τα οποία εφάρμοσε προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι πρόκειται για μια κίνηση από πλευρά κυβέρνηση η οποία είναι απολύτω αδιαφανή, η οποία είναι απολύτω ατεκμηρίωτη, η οποία είναι απολύτω αφαίρετη, δεν στηρίζεται πουθενά. Και αυτό το οποίο ζητάμε εμεί, τα ελληνικά πανεπιστήμια, επιμόνω εδώ και τρει εβδομάδε, είναι να δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση τη μέθοδο τη αξιολόγηση την οποία εφάρμοσε και η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό. Και το λέμε αυτό διότι είμαστε πεπισμένοι ότι οποιαδήποτε μέθοδο αξιολόγηση των δομών των πανεπιστημίων στη χώρα μα και αν εφαρμόσει κανεί, το αποτέλεσμα το οποίο θα βγάλει δεν μπορεί να είναι μακριά από την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ουραγή στην αναλογία διοικητικού προσωπικού, αναδιδακτικό προσωπικό ή διοικητικού προσωπικού αναφοιτητέ. Ενδεικτικά σα αναφέρω ότι ο μέσο όρο των 22 πανεπιστημίων για την αναλογία διοικητικών υπαλλήλων ανά 100 φοιτητέ στην Ελλάδα είναι 3,6 την ίδια στιγμή, σύμφωνα με, τη Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, η αναλογία στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι κατά μέσο όρο 11,5 υπάλληλοι ανά 100 φοιτητέ. 3,6 είναι στην Ελλάδα, 11,5 είναι στα γερμανικά πανεπιστήμια. Στη Μεγάλη Βρετανία, το Cambridge, για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο του Cambridge, έχει 16 διοικητικού υπαλλήλου ανά 100 φοιτητέ. Το University College London έχει 40 υπαλλήλου ανά 100 φοιτητέ. Στο Imperial College του Λονδίνου είναι 55 διοικητικοί υπάλληλοι ανά 100 φοιτητέ. Αντιλαμβάνεται κανεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολλέ τάξει στη δυσμενέστερη, σε, σε, χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρίσκονται τα ευρωπαϊκά και βεβαίως πολύ περισσότερο και τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν δεν είναι ηλίου φαϊνότερον ότι οποιαδήποτε μέθοδο αξιολόγηση των διοικητικών δομών ενός πανεπιστημίου και αν εφαρμόσει, δεν μπορεί να βγάλει κάτι διαφορετικό από αυτό που τα διεθνή δεδομένα λένε. Ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει πάρα πολύ λίγο προσωπικό σε σχέση με τις πραγματικές τη ανάγκες όπως αυτές τουλάχιστον καθορίζονται από το πλήθος των φοιτητών και εδώ να σημειώσω και έχει σημασία αυτό μιλάμε για ενεργούς φοιτητές και όχι για το σύλλο το σύνολο των εγγεγραμμένων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται και ω αιώνιοι συχνά από το Υπουργείο Παιδεία. Μιλάμε λοιπόν για του ενεργού φοιτητέ των πανεπιστημίων. Η απόλυση λοιπόν, διότι ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται των 1.400 περίπου διοικητικών υπαλλήλων, θα διαλύσει στην πραγματικότητα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό δηλαδή το οποίο θα συμβεί είναι θα έχουμε βιβλιοθήκε και δεν θα έχουμε βιβλιοθηκονόμου. Θα έχουμε γραμματείε και δεν θα έχουμε γραμματεί. Θα έχουμε εργαστήρια και δεν θα έχουμε τεχνικό προσωπικό να υποστηρίξουν τι πειραματικέ διατάξει και τι εργαστηριακέ διατάξει. Θα έχουμε φοιτητικέ αιστείε και δεν θα έχουμε υποστηρικτικό προσωπικό προκειμένου να υποστηρίζει την, τη διαβίωση των παιδιών. Ε, Γενικώ θα υπάρχουν οι υποδομέ και δεν θα υπάρχουν οι υπηρεσίε πλέον, διότι δεν θα υπάρχει το διοικητικό εκείνο προσωπικό, το ελάχιστο εκείνο διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα χρειάζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει τι ανάγκε των υπηρεσιών αυτών. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για, την πολιτική της διαθεσιμότητας. Δεν είμαστε εναντίον της, της πολιτικής της κινητικότητας γενικώ, ως μιας πολιτικής η οποία αφού αποδείξει με μια μελέτη αξιολόγησης των διοικητικών δομών πού πλεονάζει προσωπικό και πού ελείπει, θα μετακινήσει προσωπικό από εκεί που περισσεύει προς τα εκεί που υπάρχουν οι ελλείψεις. Αυτό είναι μια πολιτική ορθολογική, την οποία δεν μπορεί κανείς βεβαίως να είναι αντίθετος, πράγματι βοηθά στη διοικητική μεταρρύθμιση. Το παράδοξο στην περίπτωση των πανεπιστημίων είναι ότι δεν υπήρξε καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι τα πανεπιστήμια είναι ανάμεσα στου φορεί εκείνου που έχουν πλεονάζον προσωπικό. Το αντίθετο συνέβη. Οι αξιολογήσει που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει ότι τα πανεπιστήμια λειτουργούν με κενά στο προσωπικό του, με ελλείψει στο προσωπικό. Άρα θα περίμενε κανεί από μια τέτοια πολιτική κινητικότητα τα πανεπιστήμια να ωφεληθούν, να πάρουν προσωπικό από εκεί δηλαδή που περισσεύει και να ενισχύσουν τι δομέ του. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι όλες οι εξωτερικές αξιολογήσεις των τμήματων και των σχολών μας, όλες οι αξιολογήσεις δηλαδή που έχουν γίνει από προσωπικό, από καθηγητές εκτός Ελλάδας, από διεθνή πανεπιστήμια, όλες αυτές και το ξέρει η ΑΔΥΠ και προκαλούμε την ΑΔΥΠ να δώσει τα στοιχεία αυτά, την ανώτατη αρχή, διασφα... την αρχή διασφάλισης τη ποιότητα τη ανώτατη εκπαίδευση. Όλε λοιπόν οι εξωτερικέ αξιολογήσει σημειώνουν ότι τα τμήματα και οι σχολέ που αξιολογήθηκαν έχουν ελληπέ διοικητικό προσωπικό. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανεί ότι εδώ δεν κατηγορεί κανεί, δεν είναι κανεί απέναντι στην πολιτική τη διαθεσιμότητα ω μια πολιτική η οποία μπορεί να αναδιαρθρώσει την, ε, τη διοίκηση στην Ελλάδα. Εδώ βρίσκεται κανεί μπροστά στην εφαρμογή μια τυφλή, οριζόντια, αυθαίρετη, ατεκμηρίωτη πολιτική, η οποία διαλύει ό,τι έχει απομείνει όρθιο στην Ελλάδα. Και τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ένα από του θεσμού που στον τέταρτο χρόνο τη οικονομική κρίση, παρά το πλήγμα το οικονομικό και του προσωπικού που έχουν δεχτεί έχουν καταφέρει και παραμένουν όρθια και διακρίνονται στο εξωτερικό και παράγουν ένα έργο υψηλή ποιότητα ακόμη. Ε, λοιπόν, διαλύεται ό,τι έχει μείνει όρθιο στην Ελλάδα και αυτό είναι αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε σήμερα εδώ στι Βρυξέλλε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό θέλουμε να σα ενημερώσουμε και αυτό το οποίο ζητούμε δεν είναι να μην εφαρμοστεί η πολιτική τη διαθεσιμότητα. Είναι να εφαρμοστεί κατόπιν μελέτη και αξιολόγηση των διοικητικών δομών των υπηρεσιών στην Ελλάδα και βεβαίω και των πανεπιστημίων και ό,τι προκύψει από μια τέτοια αξιολόγηση, από μια τέτοια επιστημονική ανάλυση, την οποία θα συναποδεχθούμε από κοινού την ελληνική κυβέρνηση, εμεί δεσμευόμαστε ότι ό,τι αποτέλεσμα προκύψει θα το σεβαστούμε. Το ίδιο όμω θα θέλαμε να κάνει και η άλλη πλευρά. Ε, νομίζω ότι έχω καλύψει ένα μεγάλο μέρο. Νομίζω ότι ο πρίτανη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και μέλο του Προεδρείου, ο Πάρη ο Τσάρτα, μπορεί να συνεχίσει και να καλύψει τα όσα κενά εγώ ενδεχομένω άφησα. κλείνοντα μόνο να πω ότι η σύνοδο των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή διεκδικεί να αρθεί, να σταματήσει, να μην εφαρμοστεί το μέτρο της διαθεσιμότητας όπως εφαρμόζεται στα πανεπιστήμια, να γίνει μια μελέτη αξιολόγηση των διοικητικών μας δομών και κατόπιν αυτού πράγματι να ωφεληθούν τα πανεπιστήμια από μια τέτοια πολιτική κινητικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χρυσόγελο και το κόμμα των Πρασίνων ε, για την ευγενική και ιδιαίτερα σημαντική για εμάς πρόσκληση στο Ευρωκοινοβουλίο. Είναι πολύ κρίσιμη η περίοδος την οποία περνάμε. Ο συνάδελφος και καλός φίλος ο κύριος Μιλόπουλος νομίζω ότι έδωσε το ουσιώδες πλαίσιο του προβλήματος. Θα μου επιτρέψετε να καταγράψω κάποιες σκέψεις πρόσθετες ε, ορισμένους μικρούς προβληματισμούς και να σας μεταφέρω και μία πολύ πρόσφατη ε, εμπειρία που υπήρξε από την προσπάθεια της Συνόδου να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα στην Ευρώπη από την περασμένη Δευτέρα που ήμουνα στη Γαλλία και ε, σε μια συνάντηση των συνόδων των Πριτάνιων διαφόρων χωρών της Ευρώπης. Οι σκέψεις βασικές είναι οι εξής. Πώς μπορεί να κινείται μια τέτοια διαδικασία όταν τα κριτήρια τα οποία ζητάμε είναι δεν μας δίνονται και τελικά κατα... ό,τι έχει δοθεί στη δημοσιότητα είναι ανεπαρκές. Δηλαδή όταν επί της ουσίας μιλάει κάποιος για την ανάγκη να μειωθεί το προσωπικό σε ένα τομέα, χωρίς ε, επίσης στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα να μπορεί ο ίδιος να δικαιολογήσει το πώς κατέληξε τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. το ζήτημα αυτό συνδέεται και με την εντυπωσιακή των τελευταίων εβδομάδων προσπάθεια να δοθεί μια διάσταση, θα έλεγα, ε, διοικητική από τη μία πλευρά και εισαγγελική από την άλλη. Είναι ε, προβληματικό γεγονός το ότι για να μπορέσουν αυτά τα στοιχεία να υπάρξουν έχουμε στην ε, περίπτωση των ελληνικών πανεπιστήμιων για πρώτη φορά ουσιαστικά παρέμβαση εισαγγελική αρχής ώστε αυτό να γίνει. Το δεύτερο ζήτημα και η δεύτερη σκέψη είναι η εξή. Σε ποιο βαθμό, και αυτό επίσης το έχουμε ζητήσει, θεωρούμε ότι δεν, δεν έχει υπάρξει, αναζητήθηκαν εναλλακτικέ λύσεις. Ε, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι μιλάμε για την πρώτη τελευταία χρονιά, ουσιαστικά την τελευταία χρονιά τυπικά, όπου έχουμε την ε, Τρόικα στην ε, Ελλάδα. Την τελευταία αυτή χρονιά έχουμε τέτοιου τύπου κινήσεις. Θυμίζω ότι όχι με βάση μια λογική εξαιρέσεων, αλλά με βάση μια λογική πρόνοιας και στα πλαίσια του μνημονίου έχουμε περιπτώσεις πολύ μεγάλων επαγγελματικών ομάδων, όπως είναι οι διπλωματικοί υπάλληλοι, όπως είναι οι διπλωμάτες, όπως είναι τα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν έχουν εμπλακεί στη διαδικασία που έχουν, έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και τις πιθανές απολύσεις ή διαθεσιμότητες. Το ίδιο τυπικά συμβαίνει και με την παιδεία. Εδώ και έξι μήνες έχει πάψει να συμβαίνει. Η παιδεία έχει αρχίσει και μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία και μιλάμε εκτός από τα πανεπιστήμια και την πρωτοβάθμια και την γιατί λοιπόν έπρεπε να μπει, ειδικά αυτή την περίοδο, όπου φτάνουμε σε ένα σημείο που αν κάτι θα έπρεπε να έχει σημασία, θα ήταν ακριβώς τα πανεπιστήμια ως αναπτυξιακός μοχλός που όλοι αναζητούν. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος. Κανένα. Οι συνάδελφοι του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Αθήνας έκαναν μια προσπάθεια να βρουν το δημοσιονομικό όφελος και χάθηκαν στα μηδενικά. 0,000 και φτάσανε σε ένα τέσσερα κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει κατ' ουσία κανένα όφελος. Είναι ουσιαστικά μια κίνηση, θα έλεγε κανείς, παραδειγματισμού, συμβολική για ποιους. Ότι υπάρχουν χώροι επαγγελματικοί που έχουν να κάνουν και με ανθρώπους οι οποίοι ασκούν κρατικό λειτουργήμα όπως είναι οι καθηγητές για να είναι και αυτοί ενήμεροι και ουσιαστικά να γνωρίζουν ότι μπορεί την επόμενη χρονιά να είναι και η δική του σειρά γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν θεωρούμε ότι τα πανεπιστήμια που θίγονται αυτή τη στιγμή, τα 8, είναι τα μόνα που θίγονται. Θεωρούμε αντίθετα ότι και τα 22 πανεπιστήμια της χώρας και πιθανότατα και τα ΤΕΗ σύντομα θα έχουν μια επόμενη σειρά σε αυτό το ζήτημα. Το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ λογικό να σκεφτεί κανείς και τι έγινε αν φύγουν κάποιοι, ένας αριθμός διοικητικών υπαλλήλων. Δεν θα ορθοποδήσουν πανεπιστήμια όπως είναι το Αθηνών με 500 και 600 αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητες ή το Πολυτεχνείο ή το Αριστοτέλειο και το Πατρόν είναι τέσσερα πανεπιστήμια τα οποία όπως και αν τα δει κανεί, είναι τέσσερις βασικοί πυλώνες της ακαδημαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας με εξαιρετικά καλό διεθνές προφίλ τα οποία αν χάσουν τόσο διοικητικό κόσμο απλώς δεν θα ορθοποδήσουν γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν, τα εργαστήριά τους, δεν μπορούν να είναι η ατμομηχανή μιας ανάπτυξης που αυτή τη στιγμή κατορθώνουν και είναι. Ο προβληματισμός μας είναι καταρχάς, αφήνω τις σκέψεις και περνώ στον προβληματισμό, ότι αυτή η κίνηση έχει ένα βαθύτατα πολιτικό χαρακτήρα και χρώμα. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι είναι μια κίνηση η οποία έχει να κάνει απλώς με διαδικασίες στα πλαίσια της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση. Θεωρούμε επίσης, και αυτό είναι το, νούμερο, το δεύτερο ζήτημα το οποίο μας προβληματίζει, ότι πλάγια αλλά με συγκεκριμένο πλέον τρόπο δίνεται ένα μήνυμα ότι η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης είναι πρώτον θυρών. Και σε τελευταία ανάλυση να επισημάνω κάτι. Εάν υποτεθεί ότι η πολιτεία ήθελε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή θέλει να συζητήσει πέραν των ορίων του συντάγματος του ελληνικού ότι πρέπει να υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια ή φορείς οι οποίοι να παρέχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από πλευρά ιδιωτικού τομέα εννοώ τι υπηρεσίε του. Α το πει. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή μέσω απαξίωση ουσιαστικά ανοίγουμε την πόρτα σε αμφιβόλου ποιότητος, τρίτης θα έλεγα ποιότητα, ιδρύματα και φορεί του ιδιωτικού τομέα. Ο, η κατάσταση αυτή μας αφορά όλους και θα σας εξηγήσω γιατί. Σε αυτή την πρόσφατη συνάντηση που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα υπήρχαν εκπρόσωποι συνόδων Πριτάνιων από το Βέλγιο, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Ισπανία, ε, από, την, ε, από την Πορτογαλία και από την Ελβετία. Κοινό κανβάς, αν θέλετε, σε αυτή τη συνάντηση που είχε να κάνει με τα προβλήματα των πανεπιστημίων ήταν το γεγονός ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις έχουμε την τελευταία διετία-τριετία μια εντυπωσιακή σε κοινά χαρακτηριστικά βίαιη προσαρμογή σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Και όταν λέω βίαιη προσαρμογή εννοώ μείωση χωρίς κριτήρια και πάλι και σε διαφορετικές χώρες του αριθμού των πανεπιστημίων, μείωση με πλάγιο πάλι τρόπο του αριθμού των πανεπιστημιακών, μείωση του προσωπικού που εργάζεται στα πανεπιστήμια, αλλά βέβαια όλα αυτά με μια τεράστια διαφορά και μια δεύτερη. Η διαφορά είναι η εξή στα ευρωπαϊκά παραδείγματα. Ότι οι σύνοδοι Πυρτάνεων σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξαν συνομιλητές του κράτους με διαφωνίες αλλά συνομιλητές είτε του Υπουργείου Παιδείας είτε του κράτους σε αυτές τις πολιτικές. Συνομιλητές με διαφωνίες αλλά συνομιλητές ξαναλέω. Στην περίπτωση της Ελλάδας κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Παρά τα επιχειρήματα τα οποία σας ανέφερε πριν ο κ. Μιλόπουλος, σαφέστατα επιχειρήματα με αριθμούς, τίποτα από αυτά δεν εισακούστηκε. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα παραδείγματα τα ευρωπαϊκά δεν έχουν, με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δική μας περίπτωση. Οι συνάδελφοι, το λέω έτσι ε, με πολύ απλά λόγια, μείναμε με το στόμα ανοιχτό όταν εξήγησα ποια είναι η κατάσταση ε, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τα δικά μας. Τα δεδομένα από τη μείωση των προπολογισμών. 50 με 60% του τακτικού προπολογισμού των πανεπιστημίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τη μείωση των μισθών και τη μείωση του προσωπικού. Το προσωπικό δεν χρειάζεται να μειωθεί μόνο μέσω απολύσεων, φεύγει. Σταδιακά έχουμε πλέον ένα ουσιώδες πρόβλημα αδυναμίας να έχουμε νεότερο προσωπικό. Κανείς πλέον στην Ελλάδα δεν θα θέλει. Πριν από τέσσερα χρόνια τα πανεπιστήμια ήταν χώρος προνομιακός για πολύ κόσμο και έτσι έπρεπε να είναι. Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια τα ελληνικά σε λίγο καιρό δεν θα έχουν ελέκτορες και επίκουρους, καθηγητές και βεβαίως επειδή φεύγει πάρα πολλοί κόσμος παίρνοντας συντάξεις νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, θα έχουμε πλέον τεράστια μείωση του προσωπικού συν την δειλή αλλά σημαντική σε ποσοστά μετανάστευση η οποία εμφανίζεται από συναδέλφους οι οποίοι σταδιακά εγκαταλείπουν τη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν προβληματίζουν και εμάς και βεβαίως επισημαίνω ξανά ότι είναι και ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω λέγοντας, μεταφέροντάς σας ένα μήνυμα το οποίο είχε την ευγενική καλοσύνη να μας στείλει ο κύριος Ζαν Πιέρ Φινάνς, ο οποίος είναι ε, εκπρόσωπος της Συνόδου των Βρυτάνιων της Γαλλίας και ε, επίσης έχει σταθερή συνεργασία εδώ στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας τις Συνόδους και ε, και άλλων χωρών λάβαμε γνώση της δραματικής κατάστασης που βιώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στο πλαίσιο της τρομερής οικονομικής κρίσης που υπομένει αυτή η χώρα. Νομίζουμε ότι η μείωση της τελέχους των πανεπιστημίων κινδυνεύει να οδηγήσει τα ελληνικά πανεπιστήμια σε μια βία επιστροφή προς τα πίσω. Ομόφωνα αναγνωρίζεται ότι οι παρεχόμενοι πόροι στα πανεπιστήμια δεν είναι δαπάνες, αλλά επενδύσεις για το μέλλον. Ουσιαστικά ένα ενεργητικό πανεπιστημιακό σύστημα είναι η απαραίτητη συνθήκη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει η νεολαία με επιτυχία τις δυσκολίε του μοντέρνου κόσμου. Αποσύροντας αυτή την ευκαιρία από την νεολαία, είναι σαν να τη στερούμε τα πλεονεκτήματα και τις δεξιότητε που θα τη επιτρέψουν να ζήσει και να εξελίξει την κοινωνία. Ξαναπιάνοντας μια φράση του καθηγητή Ζαν Μαρκ Ραπ, επενδύοντας κατά τη διάρκεια της κρίσης, επενδύουμε ενάντια στην κρίση. Και ολοκληρώνοντα το επιχείρημα με το να μην στηρίζουμε την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα αποδεχόμαστε και αρνούμαστε και επιμακρών κάθε ελπίδα που επιτρέπει στις νέες γενιές να προχωρούν σε αυτό το νέο κόσμο. Παρά τις σοβαρέ δυσκολίε που γνωρίζουν, πολλέ <coughs> πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πλειοψηφικά η ανώτατη εκπαίδευση και η έρευνα είναι προστατευόμενοι τομείς η στέρηση διοικητικού και τεχνικού προσωπικού από τα ελληνικά πανεπιστήμια κινδυνεύει να τα οδηγήσει σε μια γενική αποδιοργάνωση και στη στάση ενό μεγάλου αριθμού πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει το παν για να μην φτάσουμε σε αυτό το άκρο. Ζαν Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω, θα δώσω το λόγο στην κυρία Καραμολέγκου, ε, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας μιλήσει λίγο για την κρίση, αλλά νομίζω ότι μιλώντας για την κρίση στα πανεπιστήμια, μιλάμε ουσιαστικά για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε λάθος πολιτικές για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Ε, πριν αρχίσω ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση ε, που μας επέτρεψε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και να έχουμε έτσι τη δυνατότητα να ενημερώσουμε για αυτά τα προβλήματα που μας απασχολούν και πιστεύουμε ότι δεν είναι προβλήματα μόνο της Ελλάδας, είναι προβλήματα όλης της Ευρώπης. με όσα παρουσίασαν εδώ οι δύο Πριτάνης πριν από μένα, ε, νομίζω ότι έχει δοθεί μια πολύ σαφή εικόνα ε, του γενικού προβλήματος, το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά πανεπιστήμια με την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας. Ε, ένα μέτρο το οποίο παρουσιάστηκε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι με πολύ βιαστικές κινήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι ε, το ελληνικό υπουργείο της παιδείας ε, ζήτησε στοιχεία από το ελληνικό πανεπιστήμιο ε, ζήτησε αξιολόγηση των δομών του του διοικητικού προσωπικού και των υπηρεσιών και σε ένα ασφικτικό πλαίσιο τα πανεπιστήμια αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε αυτή την ε, ανάγκη παρουσίασης αυτών των στοιχείων. Ε, τα στοιχεία παρουσιάστηκαν, αλλά έδειξαν ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν αυτή τη στιγμή έλλειμμα σε διοικητικό προσωπικό και δεν ήταν αυτό κάτι καινούριο. Ήταν κάτι το οποίο εδώ και χρόνια ε, δημοσιοποιούν κυρίως μέσω των ε, αξιολογήσεων των ε, ε, τμήματων και των σχολών που έγιναν και με διεθνείς προδιαγραφές και από ξένους και φάνηκε εκεί ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη προσωπικού. νομίζω ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι τα δύο πανεπιστήμια, δύο από τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια στα οποία πραγματικά ε, και με μόνο το άκουσμα φαίνεται πόσο φοβερή είναι αυτή η απέτηση ε, να χάσουν ε, σχεδόν το μισό προσωπικό τους. Λέμε ότι αυτή η μείωση φτάνει στην τάξη του 40 περίπου της 100, όμως στην ουσία είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί με κάποιες εξαιρέσεις που έχει κάνει το Υπουργείο στο θέμα των κατηγοριών από τις οποίες φεύγει προσωπικό, το προσωπικό που θα φύγει θα είναι από την καρδιά της διοίκησης, από την καρδιά αυτού του μοχλού στα πανεπιστήμια που ε, συγκρατεί και στηρίζει ε, την έρευνα, την εκπαίδευση ε, και πάρα πολύ σοβαρές υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές μας. Όταν μιλούμε για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλούμε για ένα τεράστιο πανεπιστήμιο το οποίο έχει 40 γραμματείες σχολών και τμήματων, έχει πάνω από 30 ε, τμήματα, 8 σχολές, ε, υποστηρίζει πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές, ε, έχει υπαίθριους χώρους, το βοτανικό κήπο, τεράστιους χώρους πρασίνου, όπου όλοι αυτοί οι χώροι χρειάζονται για τη στήριξή τους ένα διοικητικό προσωπικό το οποίο είναι απαραίτητο θα δούμε σε λίγο ότι εάν το μέτρο αυτό εφαρμοστεί, οι γραμματείες των σχολών και των τμήματων δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Ε, στις βιβλιοθήκες θα μειωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών ε, και κάτι το οποίο ε, θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, θα έχουμε μια τεράστια υποβάθμιση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, τις διεθνείς, οι οποίες είναι πάρα πολλές και ακόμη περισσότερες είναι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τα επιστημονικά προγράμματα που υποστηρίζει και στα οποία συμμετέχει αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο. Έχουμε εδώ έναν κατάλογο αυτών των προγραμμάτων. Είναι πολύ σοβαρά και μεγάλα προγράμματα ε, τα οποία όπως καταλαβαίνετε θα έχουν επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη αν δεν μπορέσουμε σωστά να τα υποστηρίξουμε και τα αφήσουμε έτσι όπως σήμερα κινδυνεύουν. Ε, επομένως ε, ε, αυτή τη στιγμή ε, το πρόβλημα ε, είναι ένα ε, διεθνές ε, πρόβλημα, το πρόβλημα των ελληνικών πανεπιστημίων. Ε, αυτό που εμείς ζητούμε, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι αφορά σε ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει και μία διεθνής, μία ευρωπαϊκή πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση να καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα στην ανώτατη παιδεία θα έχουν επιπτώσεις στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη αλλά ε, και στην ίδια την Ευρώπη. Ε, επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που ζητούμε ε, είναι ακριβώς να σταματήσει ε, αυτή η προσπάθεια υποβάθμιση, και υπονόμευση των ελληνικών πανεπιστημίων. Ε, ζητούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει αυτή την ε, υπουργική απόφαση με την οποία κανονίζονται αυτά τα θέματα της διαθεσιμότητας και σε έναν πραγματικό διάλογο με τα πανεπιστήμια, πραγματικό, όχι προσχηματικό, ε, να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία ανακύπτουν ε, αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω ότι με τρόπους αυταρχικούς και με αποφάσεις οι οποίες δείχνουν ότι δεν έχουν ληφθεί με σοβαρότητα, γιατί παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό ακόμη και αυτή η υπουργική απόφαση να αλλάζει μέσα σε δύο εβδομάδες να ε, εισάγει άλλα στοιχεία, να αναιρεί ε, προηγούμενα ή με τον τρόπο αυτό το να βρίσκονται πρόχειρες λύσεις για το πώς θα υποβάλουν τα πανεπιστήμια ε, τα στοιχεία κτλ. δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχει σχεδιαστεί ε, ε, με σοβαρότητα. Επομένως δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτές τις πρακτικές και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτό τον τρόπο ε, στις σχέσεις μας με το Υπουργείο. Ε, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή, να δούμε σοβαρά τι πρέπει να γίνει και μόνο έτσι ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι διοικητικοί υπάλληλοι των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και πολλά μέλη ΔΕΠ βρίσκονται ήδη στην έκτη εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ε, προειδοποίηση για το ότι τη δεύτερη μέρα της εφαρμογής αυτών των μέτρων τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν θα μπορούν να λειτουργούν ε, όχι μόνο με την ποιότητα την οποία είχαν μέχρι τώρα και η οποία ήταν πολύ υψηλή, αλλά θα χάσουν και τη δυνατότητα στοιχειωδών ε, λειτουργιών τους. Γι' αυτό αυτό το θέμα πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Ε, το επίπεδο και την έρευνα των ελληνικών πανεπιστημίων δεν πρέπει να την καταδικάσουμε ε, και πρέπει όλοι μαζί να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και του διερμηνεί. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρεμπέκα Χάρμ. Ε, μια σύντομη παρέμβαση και μετά ορισμένε ερωτήσεις. Ναι, καταρχά ε, ζητώ συγγνώμη που άργησα να έρθω. Ε, δεν καθυστερώ συνήθω, αλλά πράγματι σήμερα το πρωί χάλασε όλο μου το πρόγραμμα του πρωινού είχα ορισμένε πληροφορίες από τον Νίκο ήδη προπαρασκευαστικές για αυτή τη συνεδρίαση και ανησυχούσα Ανησυχούσα ιδιαίτερα για τις νέες αυτές πληροφορίες που έλαβα από την Ελλάδα, διότι κατά τη γνώμη μου εδώ γίνεται μία μεταρρύθμιση ολόκληρου του ελληνικού κράτους. Από τότε που αρχίσαμε και μιλάμε για την κρίση. Ένα κράτος που λειτουργεί, φαίνεται, κρίνεται από τους δημόσιους φορείς, από τους δημόσιους οργανισμούς και τα ιδρύματα, διότι ο δημόσιος τομέας είναι αυτός που συνδέει τους πολίτες με το κράτος τους. Αυτό το οποίο ε, βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα είναι ένα αποκλειστικά μονόπλευρο πρόγραμμα λιτότητος ε, το οποίο οδηγεί στην κατάρρευση των δημοσίων ιδρυμάτων και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Είναι η άποψη της ομάδας μου εδώ και πολύ καιρό. Ε, πολλές φορές και εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε εκφράσει τη γνώμη μας ότι αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να ε, συγχέεται με την ουσιαστική μεταρρύθμιση. Δηλαδή, ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν σημαίνει μονόπλευρη λιτότητα. Εδώ μπορούμε να επιβάλλουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση με μέσα τα οποία και, με έναν τρόπο που ούτε καν συζητιέται εδώ στις Βρυξέλλες. Πρέπει να ενισχύσουμε τα παιδαγωγικά ιδρύματα στην, Ελλάδα και αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα να γίνονται μας ενισχύουν ακόμα περισσότερο από τη, ε, ε, τα τελευταία χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα είχα μία συνάντηση με, σχολικ, με εκπροσώπους του σχολικού τομέα και βλέπω με μεγάλη ανησυχία ότι ακόμα και τα σχολεία, ε, η πρωτοβάσιμη εκπαίδευση πλήττεται και βρίσκεται σε περίοδο κρίσης. Αν αυτή η ζημιά συνεχιστεί και επαυξηθεί και εκφραστεί ξεσπάσει μάλλον και στα τριτοβάθμια ιδρύματα, τι θα γίνει με την όλη παιδεία στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ο στόχος μας είναι η καλή παιδεία, η καλή μόρφωση ε, σε όλες τις βαθμίδες τις παιδαγωγικές. Πιστεύω ότι το μέλλον είναι ζωφερό, ζωφερό, διότι αυτή η ας πούμε ελίτ του πνεύματος μεταναστεύει, φεύγει άρον-άρον από τη χώρα και πηγαίνει προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή όπου βρει ε, θέσεις εργασίας. Άρα δηλαδή το όλο θέμα της κατάρτισης, εκπαίδευση, κατάρτιση, παιδαγωγική διακυβεύεται πλέον στην Ελλάδα. Κινδυνεύει ουσιαστικά και εμείς ως πράσινοι πιστεύουμε ότι η εφαρμογή της λεγόμενης λιτότητας στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να συνεχιστεί και θα ε, κάνουμε ό,τι γίνεται για να εγκριθούν καινούργια προγράμματα και να ενισχυθούν με τα απαραίτητα κονδύλια. Όμως δυστυχώς πρέπει να πω ότι μέσα σε αυτό το σώμα εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν εκπροσωπούμε την πλειοψηφία στη Γερμανία οι σοσιαλδημοκράτες θα προσπαθήσουν να περάσουν τις θέσεις τους με τη, υπό την αιγίδα του Μάρτιν Σούλτς έτσι ώστε αυτές οι διαβουλεύσεις που γίνονται τώρα για τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία να ξεκαθαρίσουν πώς θα συνεχιστεί η μεταρρύθμιση αυτή στην Ελλάδα. Θα πιέσουν να εκφραστεί ο νέος ή όποτε γίνει αυτός κυβερνητικό συνασπισμό τη θέση για την Ελλάδα. Στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκή Υπόθεση αφορά την ελληνική κοινωνία αλλά αφορά και την Ευρώπη και του ευρωπαϊκού θεσμού. Θυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τα μέτρα δημοσιονομική προσαρμογή να μην πλήττουν το χώρο τη παιδεία, αλλά είναι λογικό η παιδεία η εκπαίδευση να είναι το εργαλείο για να βγεις από μια κρίση, για να οργανωθείς καλύτερα να προχωρήσεις μπροστά, να αντιμετωπίσεις τα λάθη σου. Επομένως είναι εντελώς παράλογη αυτή η πολιτική που πλήττει ακριβώς εκείνο το μέσο, εκείνο το εργαλείο που θα σε βοηθήσει να βγεις από την κρίση. Να θυμίσουμε ότι πέρα από τα διοικητικά θέματα και τιμή του προπολογισμού υπάρχουν 750 εκλεγμένοι καθηγητές, οι οποίοι δεν έχουν διοριστεί παρόλο ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια και ότι η Ελλάδα χάνει ε, εκπαιδευμένους, χάνει ανθρώπους στους οποίους έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και πηγαίνουν και ενισχύουν άλλες κοινωνίες και άλλες οικονομίες. Είναι εντελώς λάθος. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε μία-δύο ερωτήσεις αν υπάρχουν ε, για να πάμε μετά στο χώρο της συζήτηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, ναι, πες. Ε, in English. Στα αγγλικά. Κάριν Πάρμ, δημοσιογράφος από το University News των Βρυξελών. Καλύψαμε ήδη την κρίση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχω όμως επιπλέον ερωτήσεις. Μπορείτε να μου δώσετε τον λόγο διδασκόντων προσφυρητές. Γιατί μιλήσαμε για τον λόγο διοικητικών προσφυρητές. Αλλά καθηγητές ή διδακτικό προσωπικό προσφυρητές πριν την κρίση και σήμερα. Επίσης, δεν κατάλαβα πότε θα υλοποιηθεί το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και στη χειρότερη περίπτωση, αν όντω υλοποιηθεί δηλαδή πότε θα γίνει και τι θα συμβεί στα δικά σας πανεπιστήμια, στο, στα πανεπιστήμια που προσωπείτε εσείς. Η αναλογία, αυτό που, το πρώτο πράγμα που ρωτήσατε, επίτηδες δεν αναφέρθηκα στην αναλογία διδακτικού προσωπικού αναδιδακτικό προσωπικό, διότι και οι δύο αυτές κατηγορίες προσωπικού είναι λιματικές. Και οι δύο αυτές κατηγορίες προσωπικού, δηλαδή σε σχέση με το σύνολο των φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων, είναι πάρα πολύ μικρές σε σχέση με τις αντίστοιχες αναλογίες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Με δύο λόγια, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ελάχιστο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό σε σχέση με το σύνολο των φοιτητών τους οποίους εκπαιδεύουν. Ε, δεν έχω στοιχεία για όλη την Ελλάδα, έχω στοιχεία όμως για το δικό μου πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, όπου η σχέση, η αναλογία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ένας διοικητικός υπάλληλο περίπου για, τρεις, ε, για τρία μέλη διδακτικού προσωπικού. Για τρεις δηλαδή καθηγητές. Ένας διοικητικός υπάλληλο εξυπηρετεί επομένως τρεις καθηγητές. Και το σύνολο των φοιτητών είναι 75.000 οι εγγεγραμμένοι και 50.000 οι ενεργοί φοιτητέ, δηλαδή οι φοιτητέ οι οποίοι βρίσκονται στον ίσιν δύο έτο των σπουδών του και οι οποίοι από το Υπουργείο θεωρούνται ω οι πραγματικοί φοιτητέ, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει α το δεχτούμε ω βάση συζήτηση ότι το σύνολο των ενεργών φοιτητών μα είναι 50.000 φοιτητέ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με 750 μέλη διοικητικού προσωπικού και 2.000 μέλη διδακτικού προσωπικού, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εκπαίδευση και έρευνα για 50.000 ενεργούς φοιτητές. Είναι, η αναλογία δηλαδή είναι συντριπτική. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε, τι πρόκειται, που μας ρωτάτε, τι πρόκειται να γίνει αν εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές, είναι μια ερώτηση την οποία εμείς ως Σύνοδος των Πριτάνων έχουμε ήδη απευθύνει προς το Υπουργείο. Το ερώτημά μας δηλαδή εδώ και πολύ καιρό είναι εάν υπάρχει ένα plan B από πλευρά Υπουργείου. Όπω γνωρίζετε, στην Ελλάδα το Υπουργείο χρηματοδοτεί και θέτει το βασικό πλαίσιο λειτουργία των πανεπιστημίων, αποφασίζει τι εισόδου του και τι εξόδου του. Το Υπουργείο είναι αυτό το οποίο διορίζει λοιπόν το προσωπικό και το Υπουργείο είναι αυτό το οποίο καθορίζει τον αριθμό των φοιτητών οι οποίοι θα εκπαιδευτούν η αυτοδιοίκηση των πανεπιστήμιων έχει να κάνει μόνο με καθαρά λειτουργικά ζητήματα και όχι με βασικέ αποφάσει όπω είναι η ε, πρόσληψη διδακτικού και διηγητικού προσωπικού ή ο αριθμό των φοιτητών. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο εμεί υποβάλαμε στο Υπουργείο είναι εάν μα απομακρύνει του 1.400 διοικητικού υπαλλήλου, ποιο είναι το επόμενο βήμα τη κυβέρνηση. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα καλύψουμε εμεί τα κενά των γραμματιών που δεν θα έχουν γραμματεί, των βιβλιοθηκών που δεν θα έχουν βιβλιοθηκονόμου, των εργαστηρίων που δεν θα έχουν τεχνικό προσωπικό κτλ. Και βέβαια ε, όσο πήρατε εσείς απάντηση, άλλο τόσο πήραμε και εμείς. Ε, να προσθέσω μόνο το εξής, ότι δεν είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, όπου τόσο τα ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή οι διοικοί των ελληνικών πανεπιστήμιων, όσο και στην περίπτωση αυτή οι εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλήλων προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Δηλαδή μια πιθανή εξέλιξη την οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα είναι ότι θα έχουμε και αποφάσει της δικαιοσύνη σχετικά με αυτό το ζήτημα. Έχουμε προσφύγει στο ανώτατο, ε, στο ανώτατο δικαστήριο της Ελλάδος, Συμβούλη Επικρατεία. Ε, πολύ σύντομα να απαντήσω κι εγώ αναφορικά προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ότι εκεί αυτή τη στιγμή πριν εφαρμοστούν τα μέτρα της διαθεσιμότητας έχουμε 1.316 ε, διοικητικούς υπαλλήλους, έχουμε 1.974 μέλη διδακτικού προσωπικού ε, και οι ενεργοί φοιτητές μας ε, εντός εισαγωγικών είναι 65.682 στην πραγματικότητα φτάνουν τους 100.000 οι πραγματικοί φοιτητές και σε αυτούς τους φοιτητές δεν υπολογίζονται υπολογίζουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και άλλες κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε για να εκπληρώσουν τις ε, ε, σπουδές τους χρειάζονται μια σοβαρή ε, και στεναρή διοικητική υποστήριξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη συνέντευξη τύπου. Θα συνεχίσουμε εμείς την ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα PHS 7C50. Όλο το υλικό που έχουν φέρει οι Πριτάνες μαζί θα, είναι, ε, θα ανέβει σε λίγο στην ιστοσελίδα ε, www.χρυσόγγελος.gr ε, και είμαστε διάθεσέ και οι Πριτάνες για οποιαδήποτε ερώτηση και διαδικτυακά. Βεβαίω, θα υπάρξει σε πολλές γλώσσες και θα μπορούσαν να απαντήσουν και διαδικτυακά, μια και τα social media δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλοί κόσμο να συμμετέχει σε αυτή τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Ευχαριστούμε πολύ. ευχαριστούμε.